με προσπάθειες για να προωθήσουμε την ε, αντιμετώπιση της ανεργίας με εγχειρήματα τα οποία εναπόκειται στο Συμβούλιο, στην Κομισιόν αλλά και το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Σε μινίστρο, la discussione è chiusa. L'ordine del giorno reca ora le dichiarazioni. Τώρα έχουν τις του Συμβουλίου και της Κομισιόν για την καταπολέμηση της ομοφιλοφιλοφοβίας στην Ευρώπη. Ο Υπουργός κ. Βάμεν έχει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κύριοι Επίτροποι, όπως ο ρατσισμός και ο σεξισμός έτσι και η ομοφιλοφωνοφοβία είναι κάτι αρνητικό για τις αξίες μας και υπονομεύει το πνεύμα ανοχής και καταστρέφει τις ζωές των θυμάτων της. Γι' αυτό σήμερα το Συμβούλιο συμβαδίζει με το Κοινοβούλιο, συμφωνεί στην καταπολέμησή της. Πρέπει να προσέχουμε συνεχώς να καταπολεμούμε την άνηση μεταχείριση. Το θέμα είναι η εφαρμογή, η άσκηση των αξιών που εμφαίνονται στην χάρτα του ΟΗΕ, στη Σύμβαση των Ανθρωπίνων Πολιτικών και άλλων δικαιωμάτων, στα θεμελιώδη δικαιώματα της Ένωσης. Δεν είναι μόνο το θέμα η σεξουαλική κατεύθυνση και ταυτότης αλλά και η ελευθερία το δικαίωμα ελεύθερου λόγου έκφρασης, πολιτικής έκφρασης κλπ. Το Συμβούλιο ως συνομοθέτης ήδη έλαβε μέτρα για την προστασία των Ευρωπαίων πολιτών κατά της άνησης μεταχείρισης η οδηγία του Συμβουλίου για ένα γενικότερο πλαίσιο ίσης μεταχείρισης είναι σημαντικό βήμα. Απαγορεύει την άνηση μεταχείριση με βάση τη θρησκεία, την ηλικία, το φύλλο και την σεξουαλική κατεύθυνση. Ήδη θεωρείται λοιπόν παράνομο οι εργοδότες να μην εργοδοτούν κάποιον απλώς και μόνο γιατί είναι ομοφιλόφιλος ή γιατί είναι ετεροφιλόφιλος. Οι Ευρωπαίοι πολίτες επίσης αναμένουν ίση μεταχείριση στο, στα σχολεία, στα ιατρία κλπ. Κανείς δεν πρέπει να υφίσταται άνηση μεταχείριση λόγω της σεξουαλικής του κατεύθυνσης ή προτίμησης. Το Συμβούλιο αυτή τη στιγμή εξετάζει μία πρόταση της Κομισιόν για μία νέα οδηγία που θα επεκτείνει το δικαίωμα της προστασίας και σε τομείς εκτός της εργασίας. Κοινωνική προστασία, υγειονομική περίθαλψη, παιδεία και πρόσβαση σε υπηρεσίες και αγαθά. Γνωρίζετε πολύ καλά όμως ότι οι διαπραγματεύσεις για την πρόταση αυτή υπήρξαν πολύ δύσκολες. Το Συμβούλιο εξέτασε, εξετάζει το κείμενο από το 2008. Πρέπει να συμφωνήσουν πρώτα όλες οι χώρες μέλη. Η δουλειά μας όμως συνεχίζεται και η Ιδανική Προεδρία θα υποβάλει μία αξιολόγηση στο Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ τον Ιούνιο. Η νομοθεσία είναι φυσικά το θεμέλιο αλλά δεν αρκεί ποτέ καθε αυτήν. Έχουμε και ένα άλλο εργαλείο στη διάθεσή μας. Η αλλαγή νοοτροπίας που είναι κάτι μακρόπνοο βέβαια. Θυμάμαι ότι πριν από πέντε χρόνια οι κοινέ αξίες Κοινοβουλίου και Συμβουλίου εκφράστηκαν το 2007 έτος ίσων ευκαιριών για όλους και έτσι θυμήσαμε στους πολίτες ότι όλοι έχουν δικαίωμα σε ίση μεταχείριση ανεξαρτήτως φίλου, έθνους και σεξουαλικής προτίμησης. Κύριοι συνάδελφοι, αυτό πρέπει, τη δουλειά πρέπει να τη συνεχίσουμε. Τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι κάτι που μας βοήθησαν να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται. Και η Ένωση επίσης θέλει να πετύχει την ίδια ισότητα και στον τομέα των εξωτερικών δράσεων. Και μια απλή ματιά στις εφημερίδες αρκεί για να μας πείσει ότι υπάρχουν ακόμη, υπάρχει ακόμη ομοφιλοφιλοφοβία στην Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην καταπολέμησή της προασπίζεται τις σεξουαλικές μειονότητες που δεν προστατεύονται επαρκώς από τους πολιτικούς και τον νόμο. Η Ένωση υπήρξε ηγέτης σε τέτοιου είδους αγώνες και αυτό πρέπει να συνεχιστεί. Είναι κοινή μας ευθύνη και του Κοινοβουλίου και της Κομισιόν και των χωρών μελών και όλων των πολιτών μας. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Η Επίτροπος Ρέντινγκ. Στις 17 Μαρτίου γιορτάσαμε την Παγκόσμια Μέρα κατά της ομοφοβίας και της, της φοβίας για τα, για τα μεταφιλικά άτομα. Θέλω να τονίσω εδώ ενώπιον των εκλεγμένων εκπροσώπων των Ευρωπαίων πολιτών ότι η ομοφοβία και η μεταφιλικοφοβία είναι απαράδεκτες παραδιάσεις της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και είναι απόλυτα ασύμβατες με τις Ένωση. Γι' αυτό η Κομισιόν είναι πλήρω προσιλωμένη στην αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων με όλες τι δυνατότητες που έχει στα χέρια τη. Ω επίτροπο για τα θεμελιώδη δικαιώματα και την αποτροπή των διακρίσεων, ο στόχο μου είναι να εξασφαλίσω ότι η αρχή τη μεταχείρισης παραμένει πάντα εν ισχύ και για όλους οι λεσβείες, οι ομοφιλόφιλοι και τα μεταφιλικά άτομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθούν να είναι θύματα αποκλεισμού, μίσους, εγκλημάτων μίσους, διακρίσεων και μυσαλλοδοξίας. Το γνωρίζουμε αυτό. Γνωρίζουμε επίσης ότι τα θεμελιώδη κείμενά μας, όπως είναι η Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, απαγορεύουν κάθε μορφή Διάκριση που να βασίζεται στον σεξουαλικό προσανατολισμό. Όπως έχει εξηγηθεί στην ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, η Κομισιόν εξασφαλίζει ότι αυτές οι αρχές την χάνουν σεβασμού σε όλες τις δράσεις τη Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τα ίδια τα κράτη-μέλη όταν εφαρμόσουν το δίκαιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση η διάκριση που βασίζεται στο σεξουαλικό προσανατολισμό είναι κάτι που απαγορεύεται και από τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως την οδηγία για την απασχόληση. Η Κομισιόν έχει κάνει μια νομοθετική πρόταση για να ε, επεκτείνει αυτή την ε, υποχρέωση και στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα, όπως είναι η παιδεία. Δυστυχώς, συμφωνώ ότι το κείμενο αυτό είναι σε αδιέξοδο στο Συμβούλιο και προσβλέπω στην έκθεση που θα μας δώσει η Προεδρία για τις προσπάθειες της να προωθήσει αυτό το κείμενο. Ένα κείμενο το οποίο δυστυχώς απαιτεί ομοφωνία στο Συμβούλιο και γι' αυτό δεν έχει ευδοκιμήσει. Είναι σαφές όμως ότι υπάρχει μια συντριπτική πλειοψηφία κρατών μελών που θέλουν να υποστηρίξουν αυτό το κείμενο όχι μονάχα έχουμε νομοθεσία για τα θέματα αυτά, αλλά επίσης και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει επανειλημμένα επικυρώσει μέσω της νομολογίας του ότι οι οδηγίες για την ισότητα των φύλων στην απασχόληση και την πρόσβαση αγαθά και υπηρεσίες επίσης απαγορεύουν οποιαδήποτε ε, διάκριση σε σχέση με αλλαγή φύλου. Από νομική άποψη λοιπόν είμαστε απόλυτα σαφείς και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σε σχέση με τα νομικά θεμέλια στον τομέα αυτό. Επιπλέον, θα πρέπει να παραμείνουμε επάγρυπνοι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραμένει επάγρυπνη. Παρακολουθεί οποιαδήποτε ερώτηση κοινοβουλευτικού χαρακτήρα που υποδεικνύει προβλήματα στην εφαρμογή αυτή τη νομοθεσία, όταν πρόκειται για θέματα τα οποία εμπίπτουν στην δικαιοδοσία της Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα εγκλήματα μίσου κατά των λεσβιών, ομοφιλοφίλων και μεταφιλικών ατόμων εξακολουθούν να είναι θέμα ανησυχία, όπω η περίπτωση η δολοφονία του Ισαντζάφη στο Βέλγιο. Αυτό είναι και ο λόγο για τον οποίο η Κομισιόν έχει ζητήσει από τον Φορέα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων να προχωρήσει σε μία έρευνα σε σχέση με τα εγκλήματα μίσους και την διάκριση εναντίον των ομοφιλοφίλων, λεσβιών και μεταφιλικών ατόμων σε όλα τα κρατη και στην Κροατία γιατί πρέπει να έχουμε τα στοιχεία. Όχι μονάχα όταν συμβαίνει κάποιο έγκλημα, αλλά για να έχουμε μια σαφή εικόνα για το πού γίνονται τα εγκλήματα αυτά για να καταλάβουμε ποιε είναι οι αναδυόμενε τάσεις στον τομέα αυτό. Εν παραλίλω, η Κομισιόν συνεχίζει τι δράσει τη για μεγαλύτερη συνειδητοποίηση τη κοινή γνώμη σε όλη την Ευρώπη για να αντιμετωπιστεί η διάκριση και να προωθηθεί η πολυμορφία και η ισότητα. Υποστηρίζουμε, όπω γνωρίζετε, φορεί τη κοινωνία των πολιτών και τι εθνικέ αρχέ, το να αντιμετωπίζουμε τι διακρίσεις για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητος φίλου. Ό,τι κάνουμε στην Ευρώπη, το κάνουμε και έξω από την Ευρώπη. Η υπηρεσία εξωτερικής δράσης είναι εν επιγνώση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει η κοινότητα των λεσβιών, ομοφιλοφίλων και μεταφιλικών ατόμων σε χώρες όπως η Ρωσία, η Ουκρανία και η Μολδαβία. Για παράδειγμα, σε χώρες όπου υπάρχει όχι μονάχα διάκριση αντική και χρήση βίας, αλλά και ποινικοποίηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταδικάσει επανειλημμένα όλα αυτά τα μέτρα και έχει ζητήσει από τις αρχές των χωρών αυτών κάθε επανάληψη να σεβαστούν τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα μεταξύ των οποίων και τις αρχές της ισότητας και της ε, αξιοπρέπειας. Η κάθε Άστον έχει καταδικάσει την ομοφοβία στην ε, πρόσφατη δήλωσή της στις 17 Μαΐου ζητώντας από τις κυβερνήσεις να εφαρμόσουν με ίσο, με ίσο τρόπο τα ανθρώπινα δικαιώματα ανεξάρτητα από τη σεξουαλική ταυτότητα των ατόμων. Κάθε φορά που πηγαίνει σε μια χώρα έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπενθυμίζει αυτές τις βασικές αρχές με στεναρό τρόπο. Κυρίες και κύριοι, ως Επίτροπος για τα θέματα δικαιοσύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα κάνω ό,τι μπορώ για να γίνουν σεβαστά αυτά τα θεμελιώδη δικαιώματα από τα οποία εδράζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μονάχα κατά τη διάρκεια της διεθνού Μέρας κατά της Ομοφοβίας, αλλά και σε όλες τις μέρες του χρόνου, γιατί το φαινόμενο τη Ομοφωνία δεν έχει θέση στην Ευρώπη. Grazie Ευχαριστούμε. Τώρα οι ομιλητέ εξ ονόματο των πολιτικών ομάδων. Πρώτα το ΕΛΚΟ, κύριο Μπουζουτήλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής. Κύριε Υπουργέ, κύριε και κύριοι, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το ΕΛΚ καταδικάζει την ομοφιλοφιλοφοβία που πρέπει να καταπολεμηθεί. Αυτό πρέπει να το λέμε σαφώς και συνεχώς και με αυτή την ευκαιρία το ξαναλέμε και αυτή την εβδομάδα. Στην Ευρώπη δεν υπάρχει χώρος για διακρίσεις οποιοδήποτε είδους. Και αυτό αφορά και την ομοφιλοφιλοφοβία. Και νωρίτερα σήμερα όλες οι πολιτικές ομάδες συνεδρίασαν για να συγγράψουν ένα κοινό ψήφισμα που να μιλάει με μια φωνή κατά της ομοφιλοφιλοφοβίας. Το ΕΛΚ λοιπόν θέλει η συζήτηση να παραμείνει στοχευμένη στο πραγματικό και ενιαίο θέμα αυτό για να μην μπερδευτούν τα πράγματα και δεν βρεθεί τελικά κοινό έδαφος. Θα θέλαμε άρα να θίξουμε τα δύο ε, ακόλουθα θέματα. Πρώτον, ότι πρέπει να μην ξεχνάμε τα όρια των δικαιοδοσιών μας, δηλαδή τι μπορούμε να κάνουμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε. Και πρέπει να σεβαστούμε την αρχή της επικουρικότητας που είναι θεμελιώδης αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σημαίνει ότι θέματα που είναι δικαιοδοσία των εθνικών κυβερνήσεων πρέπει να παραμείνουν τέτοια. Δεύτερον, πρέπει να αποφύγουμε την καταδίκη μεμονωμένων χωρών ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου δεν φταίει η κυβέρνηση μιας χώρας για ορισμένες πρωτοβουλίες οι επιθέσεις. Η ομοφιλοφιλοφοβία κυρία Πρόεδρε είναι κάτι απαράδεκτο και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα καταπολεμηθεί, θα εκκριζωθεί από την Ένωση και από ολόκληρο τον κόσμο. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να γίνει αξιόπιστα και να κάνουμε σοβαρές και όχι συναισθηματικές δηλώσεις σεβόμενοι ακριβώς τα όρια των δικαιοδοσιών μας και κυρίως να μιλήσουμε όλοι με μια φωνή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για τους σοσιαλιστάς ο κύριος Κάσμαν για δυόμιση λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ χαιρετίζω τη συμβολή του κύριου Μπούσουτιλ σε αυτή τη συζήτηση. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε όλοι ως σύνολο κοινοβούλιο να καταδικάσουμε με το ψήφισμά μας την ομοφοβία η οποία σκιάζει και καταστρέφει ζωές και αυτόν που είναι η αυτοί που έχουν ομοφοβία και αυτούς οι οποίοι πλήγονται από αυτές. Τα εγκλήματα που προέρχονται από την ομοφοβία όλο και περισσότερο ε, εμφανίζονται στην Ευρώπη. Το γεγονός ότι σκοτώθηκε κάποιος στις Βρυξέλλες, όπω είπε η κυρία Επίτροπο, επειδή απλώ ήταν ομοφυλόφιλο. Η νομοθεσία της Μολδαβίας, Ουκρανία και τη Ρωσία, που είναι ένα οπισθοδρομικό βήμα. Αντί να γίνεται αποδεκτή και να είναι λόγος χαράς η πολυμορφία των ανθρώπων αντί να έχει την προστασία των κρατικών αρχών είναι υποχρεωμένοι όλοι να συμμορφώνονται με ένα πάρα πολύ στενό στερεότυπο. Δεν έχει νόημα, κυρία ε, Πρόεδρε. Έχουμε διοδίδυμους που, που γεννήθηκαν συγχρόνως. Η μία είναι ομοφιλόφιλη και η άλλη ετεροφιλόφιλη. Και για το λόγο αυτό το παιδί το οποίο είναι αγαπημένο από τους γονείς του δεν έχει πια την υποστήριξη του κράτους. Ακόμα και σε επίπεδο εκπαίδευσης που τους λέει ναι βεβαίως μπορείτε να είσαστε όποιοι θέλετε να είσαστε. Και έχουμε ιστορικά παραδείγματα ανθρώπων που έχουν σταθεί διαφορετικοί. Έχουμε ευρωβουλευτές, έχουμε πρωθυπουργούς, έχουμε προέδρους. Όχι, θέλουμε να στραγγαλίσουμε τα άτομα με την καταπίεση και τους αφαιρούμε την πληροφορία, τους αφαιρούμε την παιδεία, όλες τις ευκαιρίες για να είναι τα μοναδικά άτομα τα οποία είναι στην πραγματικότητα και τα άτομα αυτά τα οποία αξίζουν να δίνουν και να παίρνουν αγάπη. Ναι, κύριε Μπούστολη, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, θα πρέπει να σεβαστούμε τα όρια των αρμοδιοτήτων μας. Αλλά δεν πρέπει να τροποποιήσουμε αυτά που έχουμε συμφωνήσει. Δεν πρέπει να σημειώσουμε τις φιλοδοξίες μας για τα άλλα κράτη-μέλη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πιστεύω ότι αν δεν κατονομάσουμε τις χώρες αυτές, αν τις κρατάμε ανώνυμες, ενθαρρύνουμε και άλλες χώρες να συμμετάσχουν με νόμους οι οποίοι οδηγούν σε μεγαλύτερη ομοφοβία και έχουν άνηση μεταχείριση των ανθρώπων επί τη βάση σεξουαλικού προσανατολισμού τους. Κυρία Πίτροπε, κυρία Πρόεδρε, Υπάρχει τουλάχιστον ένα άτομο σε αυτή την ε, ολομέλεια που έχει υποστεί τις συνέπειες της ομοφοβίας και εγώ ως ομοφιλόφιλος άνδρας έχω αντιμετωπίσει αυτές τις συνέπειες. Εγώ όμως είχα την ευκαιρία να έχω μια οικογένεια και μια κοινωνία και να έχω παιδεία που με υποστήριξαν για να είμαι αυτό που είμαι σήμερα και να είμαι υπερήφανος για αυτό το οποίο είμαι. Είχα την ευκαιρία λοιπόν και τη φιλοδοξία που πρέπει να δοθεί σε όλα τα άτομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επέκεινα αυτή. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την ε, φιλελεύθερη ομάδα κυρία Ιντβελτ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Διαρωτόμουν για το προηγούμενο θέμα που ήταν η κρίση της Ευρωζώνης και η δημιουργία του μηχανισμού σταθεροποίησης, σταθερότητας και το Ταμείο Διάσωσης. να δεν θα έπρεπε να υπάρξει μια τέτοια δυνατότητα για αυτούς τους ανθρώπους. Είναι 5-10% του ευρωπαϊκού πληθυσμού. Συνεισφέρουν στην οικονομία μας. Συνεισφέρουν στο Ταμείο Διάσωσης για την διάσωση χωρών στις Ευρωζώνης και παρόλα αυτά δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα όπως οι άλλοι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας ούτε από τις κυβερνήσεις τους. Δεν θα πρέπει λοιπόν να ζητούμε να πληρώνουν τα ίδια, να καταβάλουν το ίδιο τέλος Ειδικά το λέω διότι αυτό δεν είναι φυσικά η λύση. Η λύση είναι να ξεκινήσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη-μέλη δίνοντας την ίδια προστασία και τα ίδια δικαιώματα σε όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι επιτέλους η χρονική στιγμή σήμερα να δράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτούς. Και είμαι υπερήφανη και με τιμά το ότι είμαι Ευρωβουλευτήνα και είμαι υπέρμαχος των δικαιωμάτων αυτών των ανθρώπων και καλοχαιρετίζω το πρώτο ψήφισμα που αφορά την ομοφοβία και κύριε Μπούσουτιλ Καλοχαιρετίζω την υποστήριξη και στην συνεργασία με την ομάδα του ΕΛΚ, διότι η διακομματική υποστήριξη για αυτό το ψήφισμα στέλνει ένα πολύ ισχυρό μήνυμα στι ίδιε τις κυβερνήσει μα, στι χώρε μα, αλλά και σε εκείνε τις κυβερνήσεις των χωρών που προαναφέρθηκαν, Ρωσίας, Μολδόβας και ποιο ήταν το άλλο κράτος. Υπάρχουν τόσα πολλά κράτη που αυτούς τους ε, πολίτες ε, με αυτή αυτές τις ιδιομορφίες τους αντιμετωπίζουν πολύ αρνητικά ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας και τα μηνύματα μίσους, οι λόγοι μίσους που εκφωνούνται από τους θρησκευτικούς και πολιτικούς ηγέτες. Όλα αυτά συνεισφέρουν στη δημιουργία ενός κλίματος μίσους αναζωπυρώνουν την μη ανοχή και την βία. Και θα ήθελα να πω και κάτι άλλο στον κύριο Μπουσουτήρ. Η διακριτική μεταχείριση δεν είναι υποχρεωτικά λιγότερο κακή από την ομοφοβία. Διότι όταν ανεχόμαστε μια τέτοια κατάσταση στέλνουμε ένα μήνυμα ότι κάποιοι άνθρωποι είναι λιγότερο ίσοι από εμάς Και αυτό δικαιολογεί την κατάσταση της ομοφοβίας. Συνάδελφοι, ζητώ από όλους να υπερψηφίσουν αυτό το ψήφισμα αύριο. Ευχαριστώ. Ενάμιση λεπτό κυρία Λούνατσεκ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε και κύριοι. Ούτε μια εβδομάδα ήταν η Διεθνή ημέρα κατά της ομοφοβίας και τη γιορτάσαμε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ένα μήνυμα σε βίντεο με παρουσία πολλών από εμά και τη κυρία Ρέντινγκ, λέγοντα στου νέου τη Ευρώπη ότι τα πράγματα βελτιώνονται. Και εγώ, ω λεσβία που έχει ζήσει σε πολύ δύσκολε εποχέ, που τουλάχιστον σε ορισμένα μέλη, μέρη αυτή τη ε, ε, Υπήρου δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα όπω είναι τώρα, ξέρω τι σημαίνει να ζει κανεί σε φόβο. Να φοβάται να περπατάει χέρι με χέρι με το αγαπημένο σου άτομο ή να το φυλάσει, να το αποχαιρετήσει σε ένα σταθμό τρένου η ομοφοβία είναι θέμα φόβου και αυτό λέει το κείμενο μας. Είναι ένας παράλογος φόβος, μια αποστροφή προς τις λεσβίες, τους ομοφιλόφιλους, τα μεταφιλικά άτομα που να βασίζεται σε προκαταλήψεις. Είναι σαν τον αντισημιτισμό και το θρησκευτικό μίσος. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το καταδικάσουμε και να εξασφαλίσουμε ότι τα άτομα δεν πρέπει να φοβούνται να ζουν τη ζωή τους πλήρως και αυτό περιλαμβάνει και μια ευτυχισμένη ερωτική ζωή. Όσο και να έχουν βελτιωθεί τα πράγματα σε πολλά μέρη τη Ευρωπαϊκή Υπήρου, υπάρχουν ακόμα λόγοι ανησυχία. Όπω αναφέρθηκε, υπάρχουν χώρε εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ρωσία, η Ουκρανία, η Μολδαβία. Υπάρχουν πολλοί, είτε οι αρχέ, είτε άλλοι που προσπαθούν να εφαρμόσουν νομοθεσία που επιτρέπουν καν να συζητάτε δημόσια το θέμα τη ομοφιλοφιλίας. Είναι τόσο σημαντικό ιδίω για του νέου οι οποίοι πρέπει να δηλώσουν δημόσια τη σεξουαλική τους ταυτότητα. Σε εμά εξαρτάται σε όλα τα επίπεδα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, να μιλήσουμε ανοιχτά κατά της ομοφοβίας, να την καταδικάσουμε, να χαράξουμε στρατηγικέ και ένα οδικό χάρτη κυρία Ρέντιν για τον αγώνα κατά της ομοφοβίας και τα ίσα δικαιώματα για του ομοφυλόφιλου και τι λεσβείε. γιατί σε αυτή την Ήπειρο θα πρέπει να καταδικαστεί η ομοφοβία και να είναι κάτι το οποίο δεν θα πρέπει κανείς μας να το υποστηρίξει για την ομάδα των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών, ο κύριος Κίρκ Κόπ, για ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, όπως είπε ο Τζορτς Βάινμπεργκ, ο, η ρίζα της ομοφοβίας είναι ο φόβος, ο φόβος και ο περισσότερος φόβος. Γιατί οι άνθρωποι αρχίζουν να φοβούνται για την, όσο οι άνθρωποι αρχίζουν να φοβούνται για την οικονομική τους ασφάλεια, δεν πρέπει αυτοί οι, φόροι, οι φόβοι να διαδοθούν και να οδηγήσουν στην απανθρωποίηση ομάδων ανθρώπων. Είναι απαραίτητο οι προσπάθειε για μια ανεκτική κοινωνία να αναστραφούν. Έχουμε όλοι διαφορετικέ απόψει σε σχέση με το ρόλο που μπορεί να παίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα θέματα αυτά. Εγώ πιστεύω ότι έχει ένα περιορισμένο ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση στην κοινωνική πολιτική, αλλά είναι μια πραγματικότητα ότι κάποιε ευρωπαϊκέ χώρε έχουν προχωρήσει πιο γρήγορα προ την ισότητα από άλλε. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι πολλέ από αυτέ ξεκίνησαν πολύ καθυστερημένα. Πιστεύω ότι είναι απαραίτητο σήμερα να είμαστε ενωμένοι για να πούμε ότι είναι μια θεμελιώδης αξία της Υπήρου μας ότι όλοι οι άνθρωποι αξίζουν μια ανθρώπινη, μια αξιοπρεπή ε, μεταχείριση ανεξάρτητα από τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό. Τίποτα λιγότερο δεν θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό από μένα κυρία Πρόεδρε. Κύριε Κύρκοπ, δέχεστε γαλάζια ή μπλε κάρτα. Ναι. Ευχαριστώ. Κύριε Κίρκοπ, συμφωνείτε ότι η συντηρητική πλειοψηφία θα έπρεπε πριν λήξει η θητεία να εγκρίνει τη, τους, το γάμο των ομοφιλοφίλων. Η απάντησή μου είναι ότι η κυβέρνηση συνασπισμού θα χρησιμοποιήσει τις σχέσεις με τρίτες χώρες για να οθήσει τα δικαιώματα των ομοφιλοφίλων διεθνώς. Και αυτή τη στιγμή κάνει διαβουλεύσεις για να εγκριθεί και ο ομοφιλόφιλος γάμος. Για την ΚΟΥΕ, ο, κύρι, κυρία ο κύριος De Κυρία Πρόεδρε, το προηγούμενο Σάββατο. Σάββατο ήμουνα σε μια συζήτηση με Ούγγρους δημοσιογράφους και πολιτικούς και κάποια κυριότερα σημεία ήταν ο νόμος για τον περιορισμό σε ετεροφιλοφιλικά μέλη μιας οικογένειας. Αυτό αφορά αυτή την ομοφοβία. Η νομοθεσία το καθιστά ανέφικτο, αδύνατο γυναίκες ε, ή για το θέμα των ομοφιλόφιλων ή για το θέμα της τρανσεξουαλικότητας να συζητεί κανείς ανοιχτά και δημόσια. Και τώρα για την υποστήριξη σε σχέση με αυτά τα άτομα θα πρέπει να υπάρξει κάποια αλλαγή με θετικά πρότυπα, με πολιτικούς που μπορούν να μιλήσουν ανοιχτά και ειλικρινά για τις σεξουαλικές τους επιλογές. Ελπίζουμε ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν βέβαια, αλλά στην πραγματικότητα τι συμβαίνει. Σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη επιδεινώθηκε η κατάσταση. Δική μας δουλειά είναι να μεριμνήσουμε, να βελτιωθούν τα πράγματα, να υποστηρίξουμε τους ανθρώπους που είναι θαραλέοι και έχουν γενναιότητα και που μπορούν να ομολογήσουν και να αναγνωρίσουν τις επιλογές τους, την κατάστασή τους και να πούν την αλήθεια για αυτήν. Κυρία Ρέντινγκ, τέτοιες κυβερνήσεις μπορούμε να στραφούμε σε αυτές μόνο όταν έχουμε θέσει σε τάξη τα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απογοητεύομαι όσον αφορά μια δυνατότητα προφορικής ερώτησης όταν αναφέρθηκε ότι δεν είσαστε λέει πρόθυμοι εσείς τώρα να συζητήσετε για μια τροποποίηση των, της αντιμετώπισης στα σχολεία αυτού του ζητήματος. Ευχαριστώ οι άλλοι εγγεγραμμένοι ομιλητές από τις πολιτικές ομάδες. Ξεκινούμε με την κυρία Στρίφλερ για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Οι πρόσφατες εξελίξεις σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες για του τους περιορισμούς στην ελευθερία του συνέρχεστε και τη έκφραση που να βασίζονται στο σεξουαλικό προσανατολισμό είναι πολύ ανησυχητικέ. Η ομοφοβία που εμφανίζεται στι χώρε Ευρωπαϊκή Ένωση και τρίτε χώρε με διάφορο τρόπο, όπω είναι βίαιη βίες δημόσιες δηλώσεις μέχρι και κλιματικές ενέργειες φόνου είναι ανησυχητικές. Υπάρχει όλο και μεγαλύτερη προπαγάνδα κατά τον ομοφιλοφίλο. Δεν μπορεί να μείνει αδρανές το όργανο μας για τα θέματα αυτά. Θα πρέπει να προσκαλέσουμε χώρες ναι, όπως η Ρωσία, η Ουκρανία, η Μολδαβία, η Λετωνία, η Λιθουανία και η Ουγγαρία να αναθεωρήσουν την νομοθεσία αυτή στο φω του διεθνού δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει. Η Κομισιόν και το Συμβούλιο θα πρέπει να λάβουν γνώση αυτών των απαγορεύσεων και να κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες μέσα στα πλαίσια του διμερούς διαλόγου και της πολιτικής εσωτερικών θεμάτων καθώς και της πολιτικής γειτονίας. Είναι λυπηρό ότι ακόμα και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα δικαιώματα των λεσβιών, ομοφιλοφίλων και των μεταφιλικών ατόμων δεν τη χάνουν πλήρου σεβασμού. Δεν μπορούμε παρά να καταδικάσουμε κάθε τέτοια μορφή διάκρισης και παρακίνησης σε μίσος και ε, εγκληματικέ ενέργειες επί βάση σεξουαλικού προσανατολισμού. Θα πρέπει όλοι να έχουν μια πρόσβαση σε θετική πληροφόρηση σε σχέση με την σεξουαλικότητά τους. Οι νόμοι αυτοί που αναφέραμε κάνουν δύσκολη και ακόμα και παράνομη αυτή την πρόσβαση σε τέτοιες πληροφορίες, κάτι το καταστροφικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο Γκυγιόμ για δύο λεπτά. Πριν από λίγες μέρες, για έβδομη συνεχή χρονιά, ε, γιορτάσαμε την ημέρα κατά της ομοφοβίας και μπορούμε να πούμε σήμερα τα πράγματα βελτιώνονται. Γιατί βέβαια παρά το γεγονός ότι έχει αποποινικοποιηθεί στις περισσότερες χώρες η ομοφιλοφιλία θα πρέπει να συνεχίσουμε να αντιμετωπίσουμε με στεναρότητα την, τις διακρίσεις κατά των ατόμων που είναι λεσβείες, ομοφιλόφιλοι και μεταφιλικά. Σε πολλές χώρες του κόσμου αυτό θεωρείται <clears throat> αξιόπινο και επίσης αξιόπινο είναι αυτό το οποίο ονομάζουν προπαγάνδα υπέρ τους, της ομοφιλοφιλίας. Το να έχει κάνει ένα προσανατολισμό διαφορετικό από το τυπικό του φίλο σημαίνει για αυτού μια αξιόπινη ενέργεια. Εμεί θέλουμε να εξασφαλίσουμε για τα άτομα τα οποία εμπλέκονται τη διεθνή προστασία. Δυστυχώ βλέπουμε στι χώρε μα ότι παραμένει ακόμα παραμένουν ελλείψεις σε νομικό επίπεδο. Είναι πολλές φορές άτομα, τα ομοφιλόφιλοι, οι οποίοι στιγματίζονται και είναι θύματα βίας οι νέοι, οι έφηβοι αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα και χρειάζεται μια προσπάθεια για να αντιμετωπιστούν τα θέματα αυτά. Είναι απαραίτητο λοιπόν να δράσουμε σε τρία επίπεδα. Πρώτα απ' όλα στην εκπαίδευση για το σεβασμό. Υπάρχουν σχολικά προγράμματα κατά των προλήψεων και προκαταλήψεων του σεξισμού και της ομοφοβίας. Επίσης, να υπάρξει δυνατότητα γάμου και υιοθεσία από ομοφυλόφιλα ζευγάρια και η νέα κυβέρνηση στη Γαλλία έχει δεσμευτεί να προχωρήσει προ την κατεύθυνση αυτή. Επίσης, να υπάρξει νομικό κολλασμό αυτών οι οποίοι κάνουν ομοφοβικές πράξει. Ευχαριστώ. Η κυρία Λάντφορτ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Με μεγάλη χαρά είδα ότι Ηνωμένο Βασίλειο είναι η καλύτερη χώρα στην Ευρώπη όσον αφορά τους ομοφιλόφιλους και αυτά τα άτομα μια και τα τελευταία χώρα τα τελευταία χρόνια οικοδομήσαμε πάνω στα θεμέλια που υπήρχαν από παλαιότερα. Δεν είναι λοιπόν ε, προς δικό μας έπαινο αποκλειστικά αυτό. Όμως σε σχέση με την κατάσταση που υπάρχει υπάρχει και μια ευρωπαϊκή διάσταση για αυτά τα άτομα. Όταν ένα ζεύγος ομοφιλόφιλων ε, που ε, ζουν, συμβιώνουν, ζουν μαζί και δεν έχουν πλέον δικαιώματα όταν μεταβαίνουν σε μια άλλη χώρα ούτε και γονεϊκά δικαιώματα. Αυτό δημιουργεί προβλήματα. Ακόμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση η αρνητική διακριτική η μεταχείριση που αντιμετωπίζουν είναι ομοφοβική και βλέπουμε ακόμα και την βία εις βάρος τους και δολοφονίες Καλωσορίζω την ε, υποστήριξη του ΕΛΚ υπό την ε, πρωτοκαθεδρία του Σάιμον Μπούσουτιλ. Η πρόοδο ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο βασίζεται σε διακομματική συνεργασία. Πριν από κάποια χρόνια είχαμε και εμείς προβλήματα σε σχέση με το, την κατηγορία, το κεφάλαιο 28 Section 28 εις βάρος αυτών των ατόμων. Τώρα όμως έχουν αλλάξει τα πράγματα. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, καταρχήν θέλω να πω στην κυρία Λάτφορντ ότι η δική μας κοινοβουλευτική ομάδα θα αποφασίσει απόψε αν το, κείμενο σύμφων, ε, την πρόταση ψηφίσματος θα την υποστηρίξει ή όχι. Ακούγοντας τη συζήτηση όμως όπως έχει διαμορφωθεί, τίνω να πω όχι, δεν θα υπερψηφίσουμε. Εγώ είμαι κατά της ομοφοβίας και είμαι υπέρμαχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όμως δεν υπάρχουν δικαιώματα ε, GPD. Αυτό είναι ανοησία. Υπάρχουν μόνο ανθρώπινα δικαιώματα. Και είναι αυτονόητο ότι για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ακόμα και για τα δικαιώματα των ομοφιλοφίλων πρέπει να αγωνιζόμαστε για να μην υφίστανται αρνητική διακριτική μεταχείριση. Γι' αυτό υπάρχει και η παράγραφος κατά της αρνητικής διακριτικής μεταχείρισης στη συνθήκη μας. Υπάρχει και η νομοθεσία κατά της αρνητικής διακριτικής μεταχείρισης και η χάρτα θεμελιωδών δικαιωμάτων. Και εκεί όπου δεν τηρούνται αυτά, αλλά τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να κατονομαστούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αυτονόητο ότι είναι αναγκαίο νομικά να δράσουμε, να αναλάβουμε πρωτοβουλίες νομικά και νομικές. Αλλά δεν συζητούμε γι' αυτό εδώ. Συζητάμε όλο το χρονικό διάστημα εδώ και πάλι σήμερα γι' αυτό για τις, ε, τους γάμους ομοφιλόφιλων. Μπορεί κανείς να είναι υπέρ ή κατά αυτών των γάμων. Όμως αυτό δεν έχει καμιά σχέση με δικαιώματα του ανθρώπου και δεν έχει καμιά σχέση και με τη χάρτα θεμελιωδών δικαιωμάτων. Στη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων αναφέρεται ρητά ότι κάθε χώρα μπορεί να αποφασίζει ελεύθερα πώς θα καθορίζει σε σχέση με ορισμούς τον γάμο και την οικογένεια. Και αυτό εντάχθηκε ρητά σε αυτή τη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ώστε να δοθεί δυνατότητα στην Ουγγαρία, στη Γερμανία και σε άλλα κράτη να πούν ότι ο γάμος είναι γάμος μεταξύ ανδρός και γυναικός. Είναι δικαίωμα αυτό που καθορίζεται σε σχέση με τη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Δεν μπορούμε να με τα πράγματα και να τα ρίχνουμε στο ίδιο καζάνι και να τα εξισώνουμε με την ομοφοβία. Μπορεί κανείς να ασκήσει επικρίσεις, αλλά σε σχέση με αυτά τα οποία είναι τρομερά και φρικτά και ισχύουν σήμερα στη Ρωσία του κυρίου Πούτιν, δεν μπορεί να τα εξισώνει όλα. Και η, κρούεται κόδωνα κινδύνου σε σχέση με τα δικαιώματα του ανθρώπου. Είναι υπερβολικά πολύτιμα αυτά για να ισοπεδώνονται και να ρίχνονται στο ίδιο καζάνι με πολιτική κοινωνική προπαγάνδα. Αυτό πρέπει να πω. Άκουσα πολλούς, ε, πολλές ε, διαμορφω... τη διαμόρφωση αυτής της συζήτησης όπως διαφοροποιούνται οι παρεμβάσεις. Είμαι κατά της ιδεολογικής προπαγάνδας παρότι δεν είμαι κατά των ομοφιλοφίλων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκούντς, 1,5 λεπτό παρακαλώ. Η κυρία Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφέρω το εξή. Και σε αυτόν τον τομέα έχουμε πάρα... Και σε αυτόν τον τομέα έχουμε πολλά να κάνουμε, διότι δεν έχουμε μια ε, μια κατεύθυνση κατά των ε, αρνητικών μεταχειρήσεων για όλους τους τομείς. Και σε σχέση με τους ε, ομοφιλόφιλους ή τα ζευγάρια ομοφιλοφιλών πρέπει να μπορούν να κινούνται ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως όταν αλλάζουν χώρα και πηγαίνουν από μια χώρα στην άλλη μπορεί να χάνουν τα δικαιώματά τους. Και η σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης προς αυτή την κατεύθυνση ε, στοχεύει. Όμως θα ήθελα να αναφερθώ στην πραγματική ελευθερία από αρνητική διακριτική μεταχείριση. Χρειαζόμαστε ένα κοινωνικό περίγυρο που θα διασφαλίζει τον σεβασμό για τους ε, διαφορετικούς ανθρώπους και την ετερότητά τους. Πολλά πρέπει να κάνουμε σε αυτόν τον τομέα. Οι πολιτικά εμπλεκόμενοι ε, όσον αφορά την παιδεία, την κατάρτιση, την εκπαίδευση, πολλά πρέπει να γίνουν. Και στην Ουγγαρία. Η Ουγγαρία θα μπορούσε να είναι ουσιαστικά υπερήφανη, διότι έχει μια μια νομοθεσία κατά της αρνητικής διακριτικής μεταχείρισης που θα μπορούσε να είναι υποδειγματική. Όμως για δεύτερη φορά συνέβη ότι η Ουγγρική αστυνομία προσπάθησε την ε, ε, εκδήλωση ε, της διαδήλωσης για την υπερηφάνεια των ομοφιλόφιλων σε μια πορεία στη Βουδαπέστη να την απαγορέψουν και να την καταστήλουν. <clears throat> Οι ομοφιλόφιλοι που θέλουν να διαδηλώσουν δεν μπορούν να διαδηλώσουν ελεύθερα βρίσκονται υπό δίωξη και αυτό συμβαίνει στην Ουγγαρία και δεν θέλουμε να συμβαίνει αυτό εκεί. Πολλά πρέπει να αλλάξουν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολλά πρέπει να κάνει. Πρέπει να διασφαλίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η υλοποίηση αυτή τη οδηγία θα πρέπει να διασφαλιστεί, θα πρέπει να υπάρξει επιτήρηση και επαγρύπνηση. Χρειαζόμαστε μια Ευρώπη χωρί αρνητική διακριτική μεταχείριση. Το Συμβούλιο θα έπρεπε την οριζόντια αυτή εγκάρσια οδηγία κατά τη αρνητική διακριτική μεταχείριση να την υποστηρίξει. Και τα κράτη-μέλη πρέπει να κάνουν πολλά για την ανοχή, ένα περιβάλλον ανεκτικότητα με διάλογο και εκπαίδευση. Ευχαριστώ. Η κυρία... Σε ευχαριστώ. Γεια Κονσάρη. Τώρα ένα λεπτό παρακαλώ. Ε, just a moment, please. Just a moment. Για στιγμή μονάχα λέει η πρόεδρος. Κυρία Γκέρνς, δέχεστε μια μπλε κάρτα. Ο κύριος Πόσελτ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Γκούντς. Γνωρίζει ότι η κυβέρνηση φίντε την ακροδεξιά, το ακροδεξιό κόμμα, το καταπολεμά με την ομοθεσία, ενώ άκουσα, διάβασα ότι σε σχέση με τους σοσιαλιστές ότι συνεργάζονται στο Κοινοβούλιο της Ουγγαρίας με τη Γιόμπικ, με το ακροδεξιό αυτό κόμμα. Αληθεύει αυτό. Θα ήθελα να μου πείτε τι συμβαίνει. Σας ευχαριστώ. Πολύ σύντομα. Όχι, δεν συμβαίνει αυτό. Δεν υπάρχει τέτοιου είδου συνεργασία στο Ουγγρικό Κοινοβούλιο. Και μάλιστα για τον εξή λόγο. Επειδή οι απόψει του Γιόμπιγκ δεν είναι αποδεκτές, είναι απαράδεκτες όχι μόνο σε αυτό το θέμα αλλά και σε όλα τα άλλα ζητήματα και θέματα. Βλέπω ακριβώς ότι η κυβέρνηση Φίντες είναι εκείνη που ακολουθεί μια κατεύθυνση ακραίων πολιτικών θέσεων και δράσεων. Διότι πολλοί πολιτικοί θέλουν οπωσδήποτε να αποφύγουν μια τέτοια ε, διαδήλωση και η αστυνομία υπό την κυβέρνηση Φίντες στην Ουγγαρία απαγόρευσε την πορεία και την ε, εκδήλωση των ομοφιλοφίλων. Δυστυχώς πολλά θα είχα να πω, αλλά δεν επαρκεί ο χρόνος. Ευχαριστώ. onorevole per un minuto. Κυρία Γιακονσάρη, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κυρία Υπουργέ, κύριε Γουάμεν, νομίζω ότι είχατε δίκιο όταν είπατε ότι η ομοφοβία είναι μια κοιλίδα στο κύρος της Ευρώπης. Εγώ όμως χαίρομαι ιδιαίτερα για την ε, ενεργητική αντιμετώπιση από την κυρία Ρέντινγκ για τα θέματα αυτά. Έχει μεγάλο κύρος η Ευρωπαϊκή Ένωση σε παγκόσμιο επίπεδο γιατί βασιζόμαστε στο κράτος δικαίου. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε όμως ότι η νομοθεσία μας παραμένει σε αυτά τα πλαίσια. Η νομοθεσία δεν πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία τα οποία οδηγούν σε διακρίσεις, ακόμα και αν είναι ε, συγκεκαλυμμένα. Δεν θα πρέπει να υπάρχει οποιαδήποτε στιγματοποίηση και αυτό είναι κάτι το οποίο θεωρούν οι νέοι ως θεμελιώδες. Ο πρόεδρος Ομπάμα στις Ηνωμένε Πολιτείε πρέπει και αυτός να τύχει επένων, όπως και ο Υπουργός Φάμεν και η Επίτροπος Ρέντιν, για τα μέτρα τα οποία ενέκρινε σε σχέση με τους γάμους ομοφιλοφίλων. Ευχαριστώ. Η κυρία Χέντ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ τα, η, τα δικαιώματα των λεσβιών, ομοφιλοφίλων και μεταφιλικών ατόμων είναι πάρα πολύ σημαντικά να τα αντιμετωπίζουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ε, είναι σημαντικό να συζητάτε το θέμα αυτό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να μείνουμε σε σύνδεση με το θέμα αυτό, γιατί κάθε μέρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνουν χώρα επιθέσεις επί τη βάση σεξουαλικού προσανατολισμού, υπάρχουν προπυλακισμοί, ακόμα και φόνοι κατά των ατόμων αυτών. Είναι πραγματικά τραγικό το 2012 στην Ευρώπη να μην έχουμε προχωρήσει περισσότερο στα θέματα αυτά. Έχουμε μια οδηγία κατά των διακρίσεων. Κάπου μαζεύει σκόνη σε κάποιο σιρτάρι τη Κομισιόν γιατί το Συμβούλιο δεν δέχεται να προωθήσει τα θέματα των ε, λεσβιών και ομοφιλοφίλων. Στην Ουγγαρία έχουμε ένα νέο σύνταγμα το οποίο λέει ότι ο γάμος είναι μια σχέση ανδρός και γυναικός μονάχα. Στη Λετωνία υπάρχει ένας νόμος ο οποίος απαγορεύει το να δίνονται πληροφορίες για την ομοφιλοφιλία. Απλές έννοιες που είναι πολύ δύσκολο να γίνουν κατανοητές. Και εκεί η μόνη λέξη που είναι κατανοητή είναι η οικογένεια. Ναι, όλοι έχουν το δικαίωμα, σχεδόν όλοι, να έχουν μια οικογένεια, αλλά όχι όλοι είναι εκτός πραγματικότητας ο ορισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την οικογένεια. Γιατί ένα από τα βασικά στοιχεία συνεργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό είναι κάτι το οποίο επηρεάζει και τα δικαιώματα των οφειλοφίλων επίσης. Ευχαριστώ. Τόμσεν για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντα ήταν επικεφαλής στον αγώνα για περισσότερη δημοκρατία και δικαιώματα του ανθρώπου και γι' αυτό αύριο θα πρέπει να εγκρίνουμε, να υπεψηφίσουμε αυτό το ψήφισμα κατά της ε, ομοφοβίας. Αυτά τα άτομα δεν πρέπει να υφίστανται αρνητική διακριτική μεταχείριση με βάση τις σεξουαλικές τους επιλογές. Όμως εξακολουθεί να ισχύει δυστυχώς το ότι αυτοί οι άνθρωποι με βάση τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό ταπεινώνονται και εξευτελίζονται παντού στην Ευρώπη. Ως πολιτικά υπεύθυνοι πρέπει να πούμε ότι αυτό πρέπει να σταματήσει και η ετερότητά τους πρέπει να αντιμετωπίζεται διαφορετικά. Πρέπει να δώσουμε μάχη κατά της αρνητικής διακριτικής μεταχείρισης. Μόνο τότε μπορούμε να περιμένουμε ότι τα δικαιώματά τους θα διευρυνθούν κοινωνικά. Και στην Δανία υπάρχει μια πρωτοβουλία όπου μπορούν να παντρεύονται και στις εκκλησίες ε, οι ομοφιλόφιλοι. Και αυτό είναι ένα βήμα απόσχησης και διαφοροποίησης όσον αφορά την ομοφοβία. Πρέπει με προοδευτικό τρόπο να δράσουμε υπέρ των αξιών και αρχών που είμαστε υπέρ αυτών στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ντέρντεν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως υπενθύμησε η κυρία Επίτροπος, το Βέλγιο είναι θλιμμένο για τη δολοφονία ενός νέου λόγω των σεξουαλικών του προτιμήσεων. Είναι ένα παράδειγμα που δείχνει δραματικά ότι είναι πραγματική η ομοφιλοφιλοφοβία και υποτιμάται ο κίνδυνος. Αυτό όμως δεν περιορίζεται στο Βέλγιο. Οι ομοφιλόφιλοι στις περισσότερες χώρες μέλη υφίστανται άνηση μεταχείριση και διακρίσει καμιά φορά και επιθέσεις. Στο Βέλγιο η κυβέρνηση εξέφρασε τη θέλησή της να εφαρμόσει νομοθεσία κατά της ομοφιλοφιλοφοβίας και των επιθέσεων κατά των ομοφιλοφίλων μιλώντας για θέματα ατομικής ελευθερίας και πρέπει όπως το Βέλγιο όλες οι χώρες να καταπολεμήσουν την ομοφιλοφιλοφοβία. Η οδηγία κατά των διακρίσεων, η οριζόντια οδηγία κατά των οδηγίων στο Συμβούλιο είναι ένα τέτοιο πρώτο βήμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Το λόγο έχουν τώρα οι ομιλητές της οφθαλμοθυρίας. Η κυρία Σίνκλερ πρώτη. Πώς θα την κάνει. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ως ένα μέλος αυτής της ομάδος ατόμων που είναι το αντικείμενο της συζήτησης, εγώ συμφωνώ με όλα αυτά που έλεγχαν εδώ, εκτός από αυτά που είπε ο κύριος Πόσελτ. Εγώ ανησυχώ όμως γιατί όλα αυτά τα μεγαλόσχημα λόγια τα οποία είπαμε κατά της ομοφοβίας είναι θετικά μεν, αλλά τα κάνουμε πραγματικότητα. Εγώ ήμουνα από τότε που είμαι μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο θύμα δύο επιθέσεων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει δράσει. Ιδίως σε τρίτες χώρες ε, υπάρχουν ακόμα περισσότερα προβλήματα. Δυστυχώς, όπως είπε και η Βαρονέσα Λάτφος, σε μια από τις χώρες που θεωρήθηκε μια από τις πιο καλές χώρες στον κόσμο για να είναι κανείς ομοφιλόφιλος, λεσβία. Δυστυχώς υπάρχουν άλλοι άνθρωποι στην, στον κόσμο που δεν μπορούν να πούν το ίδιο και γίνεται τώρα στην Ουκρανία ένα ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα το Ευρώ που έχει σαν ε, συνδιοργανωτή την Πολωνία και δυστυχώς πολλοί από εμά. Θα πρέπει να μεταβούμε στην Ουκρανία. Ε, όπως ξέρετε σήμερα το Υπουργείο Εξωτερικών έχει κάνει μια προειδοποίηση για τους ανθρώπους, δηλαδή σαν ταξιδιωτική οδηγία να είναι πολύ προσεκτικοί όταν μεταβαίνουν στην Ουκρανία. Δεν θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μποϊκοτάρει αυτό το πρωτάθλημα αν δεν μπορούμε να προστατεύσουμε τους πολίτες. Ευχαριστούμε. Μοργάντη. Πολύ σωστό να καταδικάζουμε κάθε μορφή βίας. Όμως υπάρχουν και σημεία τα οποία δεν μπορούμε παρά να λάβουμε υπόψη. Καταρχήν η οικογένεια που απαρτίζεται από, άντρα από έναν άντρα και μία γυναίκα για να γεννηθούν παιδιά που δεν μπορούν να γεννηθούν από το ίδιο φύλλο. Μπορούν να συζούν αν θέλουν οι ομοφιλόφιλοι, αλλά δεν μπορούμε να μιλήσουμε για γάμο, δεν μπορούμε να μιλάμε για γάμο και για υιοθεσία. Δεν μπορούμε να κινούμαστε κατά φύσης. Όλα τα άλλα αποτελούν στήρο εγωισμό που φτάνουν σε επιπολαιότητες όπως το να μιλάμε για άνδρες μητέρες. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τη φυσική ροή των πραγμάτων. Φλασίκοβα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ, ε, κυρία Επίτροπε, ε, κυρία Πρόεδρε. Δεν θα μιλήσω για χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, όπου, διότι υπάρχει πρόβλημα με την ομοφοβία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση την περασμένη εβδομάδα ένα μέλος ε, του Κοινοβουλίου, ένας βουλευτής του Κοινοβουλίου της Σλοβακίας είπε ότι οι άνθρωποι αυτοί θα έπρεπε είτε να εγκλειστούν είτε να θεραπευτούν. Άρα δεν μιλάμε μόνο για εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως αλλά και για εντός. Και όταν κάτι τέτοιο συζητιέται ε, δεν ρωτάω ποιες είναι οι σεξουαλικές τους ε, προτιμήσεις θέλω να έχω φίλους, φίλους με τους οποίους μπορώ να βασιστώ που έχουν τις ίδιες προοπτικές και τις ίδιες απόψεις για τη ζωή. Γι' αυτό και λυπούμε ότι ε, φυστάμεθα τέτοιες ε, ε, επιθέσεις όχι μόνο από τον χώρο εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως αλλά ακόμη και από τους πολιτικούς εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Εάν λοιπόν δεν μπορεί να υπάρξει νομοθεσία στα διάφορα κράτη-μέλη, ίσως το Ευρωπαϊκό η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να νομοθετήσει διότι δεν μπορεί κανείς να αφήσει τα θέματα αυτά αποκλειστικά στα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Η κυρία Πρέντεργκαστ. Thank you, uh, uh, χρόνια και χρόνια καταγγέλνουμε την αποφοβία και τις ενέργειες από άτομα και αναπτύσσονται ε, τέτοιες ε, τάσεις ακόμη και στις γειτονικέ χώρες αλλά και στα κράτη-μέλη. Ε, σε μια ομάδα που συνεδρίασε είχα την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας Επίτροπε Ρέντινγκ και με εκπροσώπους από το Συμβούλιο και ε, υποσχεθήκαμε στις αδελφές μας ότι θα βελτιώσουμε τα πράγματα. Όπως σωστά ανέφερε το Συμβούλιο, οι διακρίσεις με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό δεν συμβαίνει μόνο στον χώρο εργασίας. Καλύπτεται αυτό από την κοινωτική νομοθεσία. Ε, θα έπρεπε να έχουμε ίση μεταχείριση άσχετα από τη θρησκεία, το φύλλο κτλ ε, των ανθρώπων, αλλά αυτό παρεμποδίζεται να προχωρήσει στο Συμβούλιο. Δεν με ενδιαφέρουν τα θέματα της επικουρικότητας. Θα ήθελα όμως να καταλάβουμε όλοι ότι πρέπει να ενισχύσουμε τη σχετική νομοθεσία. Ο κύριος Κορνέλησεν τώρα. Η κυρία Κορνέλησεν, με συγχωρείτε. Την Κυριακή ήμουνα στην Ουκρανία. Στην Ουκρανία είχα ελπίσει να συμμετάσχω στην ε, πρώτη παρέλαση των γκέι, των ομοφιλοφίλων. Δυστυχώς όμως χρειάστηκε να ακυρωθεί γιατί περισσότεροι από 500 εθνικιστές απειλούσαν και η αστυνομία δεν φαινόταν να είναι ικανή να προστατεύσει την παρέλαση τουλάχιστον δεν ήθελε. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο νομοσχέδια στην Ουκρανία τα οποία ουσιαστικά θα δυσχεράνουν ακόμη περισσότερο την ζωή για τους ομοφιλόφιλους και τις λεσβίες. Είναι ευρωπαϊκή χώρα αυτή, θέλει διασυνδέσεις με την Ευρώπη, θέλει ελεύθερο χώρο εμπορίου και θα ήθελα να ζητήσω από την Επικομισιό να το καταστήσει σαφές ότι το ελεύθερο εμπόριο και η ελεύθερη κυκλοφορία ανθρώπων μπορεί να συμβεί. Μπορούν να συμβούν μόνο όταν υπάρχει απόλυτη σεξουαλική ελευθερία. Συνάδελφος Μιράντα τώρα. Ευχαριστώ. Κυρία Επίτροπε, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η πρόταση εφαρμογής της οδηγίας κατά των διακρίσεων και θα πρέπει να την ε, ξεμπλοκάρουμε κατά κάποιο τρόπο. Νομίζω ότι θα πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν ε, βουλευτές που καταπολεμούν την ε, φυσική βία, τη λεκτική βία, τις ε, εκδιώξεις, τις απολύσεις, την ε, έλλειψη ελευθερίας και τη μη σωστή αντιμετώπιση των ανθρώπων, διότι κάθε μέρα γίνονται πράξεις κατά των ομοφιλοφίλων και καταδικάζονται και σε θάνατο. Γι' αυτό θα πρέπει να εγγυηθούμε τα δικαιώματα και να θα πολεμήσουμε τις διακρίσεις κατά των λεσβιών, ομοφιλοφίλων, αμφιφιλοφίλων και ούτω καθεξής. Ευχαριστώ. Η Επίτροπος Ρέντινγκ έχει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, <clears throat> νομίζω ότι υπήρξε σχεδόν ομοφωνία μεταξύ των ομιλητών ότι η ε, ομοφοβία δεν έχει θέση στην Ευρώπη ούτε ε, και καλυμμένα ούτε εκδήλως και ε, ούτε στα κράτη που είναι μέλη εδώ και καιρό και στα νέα κράτη-μέλη εναντίον οποιοδήποτε πολίτη ασχέτως του οποίου είναι ε, εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στις χώρες που θέλουν να έχουν σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το είπα σαφώς στην ομιλία μου και αναφέρθηκα στην κυρία Άστον η οποία τακτικά επεμβαίνει σε συγκεκριμένα θέματα ε, στα κράτη αυτά περί των οποίων ομιλούμε. Επειδή όμως συμφωνώ με όλα ε, κύριε Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε δεν θα αναφερθώ σε όλα τα θέματα αλλά μόνο μόνο σε ένα το οποίο έχω απαντήσει γραπτός επανειλημμένος και ήταν σκόπιμο να απαντήσω και εντός του Κοινοβουλίου για να διευκρινίσω τη θέση μου. Είναι η σχέση μεταξύ την οδηγία ελεύθερης διακίνησης και την αμοιβαία αναγνώριση των ζευγαριών ιδίου φίλου, διότι ξέρετε ότι προβλέπεται η ε, εγκατάσταση ασχέτως της αναγνωρίσεως των γάμων μεταξύ μελών του ιδίου φύλου και ε, στο άρθρο 24 της οδηγίας αυτής λέγεται ότι τα ζευγάρια ιδίου φύλου που εξασκούν το δικαίωμα ελεύθερης διακίνησης έχουν τα ίδια δικαιώματα όπως ε, τα τα ε, παρόμοια ζευγάρια ή τα ε, κράτη υποδοχής. Δεν σημαίνει ότι θα αποκτήσουν με περισσότερο, ε, περισσότερα δικαιώματα στα κράτη-μέλη από ό,τι εξασφαλίζονται τους πολίτες των κρατών μελών. Και το θέμα της αναγνώρισης των γάμων δεν υπησέρχεται στην εφαρμογή αυτής της οδηγίας και για να εφαρμοστεί σωστά τα κράτη-μέλη δεν χρειάζεται να αναφερθούν στην αναγνώριση αυτών των ενώσεων αλλά απλώς να χορηγήσουν δικαίωμα εισόδου και παραμονής στα ζευγάρια αυτά και στα μέλη της οικογενείας τους περιλαμβάνοντας τους συντρόφους και ε, του συζύγους ασχέτως του σεξουαλικού προσανατολισμού δηλαδή είναι υποχρεωμένοι να δεχθούν το σύζυγο του πολίτη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ασχέτως του προσανατολισμού αλλά χωρίς να είναι υποχρεωμένο στο κράτος υποδοχής να αναγνωρίσει το γάμο αυτό. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει αυτή η αναγνώριση τι πρέπει να κάνουμε και θα αναφέρω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Υπήρξε η απόρριψη των πολωνικών αρχών να χορηγήσουν ένα ε, ε, ε, ένα πιστοποιητικό για να μπορέσουν να συζευχθούν δύο μέλη του ιδίου φίλου και ε, σαν Ευρωπαϊκή Ένωση είπαμε ότι αυτό δεν συνάδει με την οικογενειακή ζωή και οι πολωνικές αρχές μας είπαν ότι θα ληφθούν μέτρα για να διαγραφεί το φίλο του ε, μελλοντικού συζύγου. Αυτό για να σας εξηγήσω τι προβλέπει ο νόμος και πώς μπορούμε χαμηλοφόνος να ε, επέμβουμε στην εφαρμογή της νομοθεσίας σε ένα κράτος μέλος κατά τρόπεν ώστε να αλλάξουν οι πρακτικές οι οποίες δεν συνάδουν με τις, ε, τη νομοθεσία και τους κανόνες κρατών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο Υπουργός Βάνεν. Καπιτά Αγαπητά μέλη του Κοινοβουλίου, κύριε Επίτροπε, αν θα πρέπει να συνοψίσω τις συνέπειες θα έπρεπε πρώτα απ' όλα να διαπιστώσω ότι μιλάμε για το Κοινοβούλιο, μιλάμε για την Κομισιόν, μιλάμε για το Συμβούλιο, αλλά τελικά όλοι βρισκόμαστε στο είδο μήκο κύματο. Δηλαδή λέμε ότι οι διακρίσει μπορούν να καταπολεμηθούν και πρέπει να προασπίσουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα. Αυτό είναι και το βάθρο, η βάση της ευρωπαϊκής συνεργασίας. Όπως είχα την ευκαιρία να το πω με σαφήνεια στη συζήτηση σήμερα, το Συμβούλιο οπωσδήποτε ακολουθεί την ίδια γραμμή με το Ευρωκοινοβούλιο. Είναι αυτονόητο ότι προστατεύουμε την αρχή σύμφωνα με την οποία κανένας πολίτης δεν πρέπει να υφίσταται διακρίσεις λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού. Αυτό είναι μια βασική αρχή. Συνεπώς, είναι ουσιώδες να υπογραμμίσουμε ότι όλα τα κράτη-μέλη πρέπει να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να επιτρέψουν σε όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά τους. Και αυτό πρέπει να γίνει και στο γράμμα και στην εφαρμογή του νόμου. Η Δανική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνεπώς, θα συνεχίσει να εργάζεται για την ε, οδηγία κατά των διακρίσεων που θα μπορούσαν να αποτελέσει μια σημαντική συμβολή ώστε να μην επιτρέπεται η διάκριση και εκτός του χώρου εργασίας. Σημείωσα όσα ελέγχθησαν και, και πολύ σωστά ελέγχθησαν εδώ σήμερα. Ε, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι θα τα αναφέρω στο Συμβούλιο. Ταυτόχρονα σας υπόσχομαι ότι η Δανική Προεδρία θα ενδιαφερθεί για την προστασία αυτών των θεμελιωδών δικαιωμάτων μέχρι και το τελευταίο λεπτό της προεσδρίας μας. Και βεβαίως θα συνεχίσουμε και μετά σαν ένα κράτος μέλος μεταξύ άλλων 27. Λοιπόν, για όλους μας, είτε είμαστε μέλη της Κομισιόν του Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, δεν έχει σημασία η θρησκεία μας, η σεξουαλικότητά μας, η προέλευσή μας, όλοι μας έχουμε ένα κοινό έργο. Πρέπει να φροντίσουμε η ομοφοβία, η οποία αποτελεί δυστυχώς κομμάτι της ιστορία μας, η ομοφοβία αυτή να μην μπορεί ποτέ πια να είναι στοιχείο του κοινού μας μέλλοντος. Αυτό είναι το έργο μας. Σας ευχαριστώ όλους. Σας ευχαριστώ και εγώ. Υπάρχουν ε, πέντε προτάσεις ψηφίσματος μετά από τη συζήτηση. Κλείνει η συζήτηση και η ψηφοφορία θα διενεργηθεί την πέμπτη. Τώρα προβλέπεται η